Ευχαριστώ, συνάδελφε, ε, πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μαμίκης, γιατί με... και τον ευχαριστώ ως κοιόδη εισηγήτρια. Ο εισηγητής εξήγησε πολύ σαφώς, πολύ συγκεκριμένα τη δουλειά που έκανε, το πρόβλημα που υπάρχει με, την με τη θέση στο εμπόριο και τη χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, λοιπόν. Θέλω να πω στα μέλη της Κομισιόν ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ότι προφανώς ε, οι πρόδρομες ουσίες συνδέονται με την καταπολέμηση της δημοκρατίας και σας στηρίζω και σας ε, παρακινώ να δουλέψετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Φυσικά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά νομίζω ότι ήταν κομβική σημασία να τροποποιήσουμε την νομοθεσία που ισχύει σήμερα για να ελέγξουμε καλύτερα την πώληση των προδρόμων ουσιών εκρηκτικών. Το ξέρουμε και το υπενθυμίσατε συνάδελφε ότι αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Το 40% περίπου, δηλαδή μία επιθέση στις δύο, οργανώνεται και προετοιμάζεται χρησιμοποιώντας τέτοιες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών. Η θέση στο εμπόριο λοιπόν στις επιγραμμικές πλατφόρμες είναι προβληματική ε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η έκθεση που μας παρουσιάσατε σε αδρές γραμμές είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας και η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα συμφωνεί με αυτά που είπατε και με τις κατευθυντήριες γραμμές που σκιαγραφίσατε και χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες σήμερα το πρωί Νομίζω ότι η τροπολογία 6 και 7 που αφορούν το άρθρο 7 για την ενημέρωση για την αλυσίδα ανεφοδιασμού, εκεί όλες οι πρόδρομες ουσίες ε, εκρηκτικών θα πρέπει να ρυθμίζονται, λέτε, και όχι μόνο οι ε, πρόδρομες ουσίες υπό περιορισμό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή γραμμή δράσης αυτή. Επίσης, ε, μιλήσατε για την αδειοδότηση, τις άδειες. Δεν αναφέρατε την τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα τα κράτη να ζητήσουν πληροφορίες συμπληρωματικέ. Ε, αυτά είναι θετικά και χρήσιμα στοιχεία για την οργάνωση της πώληση και τις θέσεις στο εμπόριο αυτών των ουσιών. Τώρα προσωπικά κάποιε απόψει. και εξ ονόματο των συναδέλφων της κοινοβουλευτική μου ομάδας θα υποβάλω κάποιε τροπολογίες, μία τροπολογία για την σαφήνεια των ορισμών καθώς και για, την, για τις προθεσμίες με τις οποίες μιλήσατε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μικρές προθεσμίες, συγκεκριμένες, ξεκάθαρες, απόλυτα, ούτω ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενδιαφερόμενες να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη χρήση. Επίσης, κάτι πολύ προφανές. Εάν υπάρχει μια ύποπτη συναλλαγή και, αυτή, και για αυτή δοθούν πληροφορίες πολύ αργά, μπορεί να έχει σοβαρότερες συνέπειες κάτι τέτοιο. Είναι θέμα χρόνου μερικές φορές. Ε, πριν από 7-8 εβδομάδες στη Γερμανία υπήρξε ένα παράδειγμα. Εντοπίσαμε πολύ γρήγορα ε, από την πλατφόρμα eBay, η οποία πλατφόρμα προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να γίνει μία ε, επίθεση και την αποτρέψαμε. Για την εφαρμογή διαδικασιών, για την ε, ενημέρωση για μια τέτοια ύποπτη συναλλαγή, μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό το θέμα, θα το κάνουμε. Επίσης, θα ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή στα θέματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης εγώ ήρθα σε επαφή με πολλούς ε, οικονομικούς φορείς ε, που δεν είναι κατά της πρόταση, αλλά διερωτώνται τι πρέπει να κάνουν, πώς θα οργανωθεί το πράγμα και πώς θα οργανωθούν οι ίδιοι. Νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των ατόμων που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι θα μας επιτρέψει, δεν είναι και εύκολο, αλλά θα μπορούσαμε όμως να μειώσουμε τα, τις που υπάρχουν στο σύστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας τακτικός και οργανωμένος διάλογος μεταξύ των αρχών και των διοκτικών αρχών συγκεκριμένα των κράτων μελών και των ελεγκτικών αρχών με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω, ώστε ο καθένας να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που, εντάχει που σας λέω, δεν τα κάλυψα όλα. Μιλάω ως όδηση εισηγήτρια και εκφράζω και τις ναι. απόψεις της κοινοβουλευτικής μου ομάδας, ευχαριστώντας ακόμα μία φορά τον εισηγητή για όλα όσα έκανε στο παρελθόν και όλα όσα θα κάνει. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ. Είστε σκιώδης εισηγήτρια για τους φιλελεύθερους. Τώρα θα δώσω το λόγο στην σκιώδη των Πρασίνων, κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι εγώ θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ θετικό το να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε σωστά τα χημικά προϊόντα και για το περιβάλλον. Για μας ε, είναι κάτι βέβαια το οποίο συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με ε, την ασφάλειά μας. Υπάρχει βέβαια το θέμα της συλλογής προσωπικών δεδομένων και η διάρκεια, ο χρόνος διατήρησης των συγκεκριμένων δεδομένων ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε αυτό το σημείο της πρότασης να καταθέσουμε τροπολογίες. Κατά τα άλλα υποστηρίζουμε την πολύ καλή δουλειά. Thank you, Mrs. Valero. Uh, colleagues, uh, we also have the Commission present. Uh, I give the floor to Deputy Director General at DG Home, Mr. Onidi. Uh, Mr. Onidi, you have three minutes. Uh, uh, Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μαμίκης και τους Σκιώδης ε, για την ταχύτατη και ποιοτική δουλειά την οποία έκαναν σε μια σημαντική πρόταση. Νομίζω ότι ο εισηγητής ε, τεκμηρίωσε την πρότασή του Έχουμε κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να κλείσουμε στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και παράλληλα με τα, μέτρα που πήραμε για τα φορητά όπλα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τις πρόδρομες ουσίες. Είναι κάτι στο οποίο έχει σταθεί επανειλημμένα ο Επίτροπος Κέγκ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, στα πλαίσια της αρμόδιας επιτροπής και περιλαμβάνεται στην έκθεσή της, την πρόταση έκθεσης της επιτροπής. Θα στηρίξουμε και τις τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται. Υπάρχουν ορισμένες προτάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά το κείμενο. Ευχαριστούμε που κρατάτε ε, το self acid στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη πρόταση. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον καθαρισμό ε, σε πισίνες, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεαστούμε ιδιαίτερα από τις πιέσεις αυτής της κατηγορίας. Θα πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να ανανεώνουμε ε, τον κατάλογο αυτό μέσω της διαδικασίας επικαιροποίησης θα έλεγα έτσι ώστε η δουλειά η οποία θα γίνεται όταν εμφανίζονται νέους ουσίες στα χέρια των τρομοκρατών να μην χρειάζεται μακρά διαδικασία για την συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσης ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που κάνατε σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις και σε σχέση με τον έλεγχο και την διαπίστευση σε εισαγωγικά των επιχειρήσεων πριν από μια συγκεκριμένη πώληση, όπως και για τα μέτρα και τις διατάξεις για τον έλεγχο και την εποπτεία. Ευχαριστούμε και για κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως η βελτιωμένη διαφάνεια, η υποχρέωση ενημέρωσης προς τους ε, εργαζομένους στην επιχείρηση, τους ενδιάμεσους πολιτές και τους αγοραστές, όπως και τα θέματα της κατάρτισης που ανάφερε και η κυρία Γκρίσμπεκ είναι σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ που αναφέρεστε και στη ΣΕΠΟΛ και σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε μέσω της υπηρεσίας αυτής. Τώρα για τις ε, δικτυακές πωλήσει γνωρίζουμε ότι και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει ενδιαφέρον έτσι ώστε να διευρυνθεί η συγκεκριμένη θα έλεγα πρόταση. Νομίζω ότι θα συμπεριληφθεί καλύτερα, θα ενταχθεί καλύτερα στην γενική πολιτική μας σε σχέση με τις διαδικτυακές πολιτικές. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ευχαριστώ τον κύριο Μαμίκινς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Συνάδελφοι, περιμένω ε, περαιτέρω καρποφόρο συνεργασία. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις από όλες τις πολιτικές ομάδες, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο σημείο 11 της σημερινής διάταξης. εξέταση σχεδίου έκθεσης για το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εδώ η κυρία Κιγκαγκάλ, που είναι η συγγήτρια. Είναι η συγγήτρια, αλλά δυστυχώς δεν είναι παρούσα. Ούτε υπάρχει κάποιος που να την αντικαθιστά. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε ένα-δύο λεπτά Μήπως και προσέλθει η κυρία Κίνγκα και θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Ευτυχώς ήρθε και η συγκήτριά μας, η κυρία Γκάλ. Έχετε λόγο. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Τόσα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Λοιπόν, για το, ταξιδετικό, το προσωρινό ταξιδετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της, ε, του, της σχετικής οδηγίας. Η Κομισιόν της 96 κάθετος 406 υπέβαλε λοιπόν αυτή την πρόταση φέτος, την παρουσίασε Το Κοινοβούλιο έχει μόνο ρόλο διαβούλευσης Συζητήσαμε και με την νομική υπηρεσία, η οποία επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτή είναι η νομική βάση. Λοιπόν, η Κομισιόν θέλει να απλοποιήσει τις τυπικές διαδικασίες για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν βρίσκονται σε τρίτες χώρες και έχουν ε, χάσει ε, το διαβατήριό τους, ή έχει καταστραφεί ή έχει κλαπεί το διαβατήριό τους. Δηλαδή όταν βρίσκονται σε κατάσταση που, βρίσκονται, που χρειάζονται βοήθεια. Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο λοιπόν θα μπορούν να το παίρνουν και από άλλε προξενικέ ή προσβεστικέ αρχέ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καινούριο αυτό. Είναι κάτι που υπήρχε και το, στην πρόταση του 1996. Ε, βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και η τρέχουσα μορφή αυτού του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από χαρακτηριστικά ασφάλειας αλλά ε, δεν προστατεύεται και παρκώς έναντι πλαστοποίησης, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που δεν εκδίδουν πλέον το ταξιδιωτικό αυτό το προσωρινό έγγραφο, ακριβώ γιατί θεωρούν ότι δεν είναι πλέον ασφαλέ. Η προταση του 1996 επίση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Συμβουλίου του 2015 για την προστασία, ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, στο ψήφισμά του 2017 για την έκθεση για την Ιθαγένεια κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, πιο ασφαλές, μια νέα πιο ασφαλή μορφή αυτού του ταξιδιωτικού εγγράφου. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το θέμα που συζητάμε. Η Κομισιόν με την ε, τρέχουσα πρότασή της λοιπόν ε, ευθυγραμμίζει το καθεστώς γύρω από αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο με τη σημερινή εποχή, ενισχύει τα χαρακτηριστικά ασφάλεια του, ε, αποτρέπει έτσι, αποτρέπεται έτσι καλύτερα η κακή χρήση ή ε, κατάχρηση αυτών των εγγράφων και νομίζω ότι όλα αυτά ε, αποβαίνουν προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή αφενός να χαίρουν προστασίας και συνδρομής από τις προξενικές αρχές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό εκτός Ένωσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και των ίδιων των πολιτών. Νομίζω ότι η πρόταση είναι καλή, πρέπει να υποστηριχθεί χωρί τροπολογίε. Χρειάζεται οι Ευρωπαίοι πολίτε όταν βρίσκονται σε τρίτε χώρε να ε, την χάνουν συνδρομή και βοήθεια από τι προξενικέ αρχέ όλων των κρατών μελών. Λοιπόν, 25 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και από εκεί πέρα θα δούμε ε, κατά πάσα πιθανότητα τις ε, τροπολογίες αυτές στις 5 Νοεμβρίου στη συνεδρίασή μα. Ευχαριστώ κυρία Γκάλ. Κυρία Κινίτσι από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κίνγκα Γκάλ, που μας παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης Μα ακούτε καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι ευχαριστώ την Πρόεδρο και την εισηγήτρια, την κυρία Κίνγκα Γκάλ, που μας παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης για την αναθεώρηση του προσωρινού εγγράφου, ταξιδιωτικού εγγράφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η εισηγήτρια, είναι ένα σημαντικό έγγραφο και πρέπει να επικαιροποιηθεί βεβαίως για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία στο εξωτερικό και για να τους επιτρέψουμε να επαναπατριστούν με, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Να πω κάτι που υπόθηκε. Το έγγραφο εξασφαλίζει το βασικό δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης σε, τους εξασφαλίζει διπλωματική και προξενική προστασία, όπως προβλέπει και το άρθρο 46 της Χάρτας και είναι μία απόδειξη της α, σημασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών τη στιγμή που ένας πολίτης της Ένωσης ε, αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αναθεώρηση της νομικής βάσης του προσωρινού εγγράφου ταξιδιού είναι, σημαντικ... είναι βασική προϋπόθεση για να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά ασφάλειά του και να μειωθεί ο κίνδυνος παραποίησης, ο, ο κίνδυνος απομίμησης, ε, παραποίησης, απομίμησης κτλ. Και να μειώσουμε τη δυνατότητα που έχουν οι εγκληματικές οργανώσεις ή οι τρομοκρατικές οργανώσεις να χρησιμοποιούν τέτοια πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα. Επίσης, ε, τα πιο υψηλά πρότυπα ασφαλείας, πιστεύω, όπως έλεγε και η συγγήτρια, θα κάνουν ε, πιο αποδεκτά τα έγγραφα αυτά σε τρίτες χώρες και θα διευκολύνουν ε, τα τις διατυπώσεις στα εξωτερικά σύνορα θα μειώσουν το κόστος και τις δυσκολίες για τους πολίτες που έχουν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση. Συνοπτικά, συμφωνώ με αυτά που είπε η συγγήτρια και γι' αυτό εγκρίνουμε την πρόταση και την υποστηρίζουμε να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες για αυτό το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο ε, που θα καλύψει πολίτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από δικές τους προξενικές διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική ομάδα και εγώ πιστεύουμε ότι η πρόταση συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερο θετική για τρεις λόγους. Πρώτον είναι μια πρόταση η οποία είναι προς το συμφέρον των πολιτών θα επιτρέψει στους πολίτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από το προξενείο της χώρας τους, οι οποίοι έχασαν το διαβατήριό τους ή εκλάπη ή καταστράφηκε, τους δίνει η δυνατότητα ή οδήποτε άλλο προξενείο της Ένωσης να τους δίνει ένα έγγραφο ταξιδιωτικό, ασφαλές, ε, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην ίδια την ασφάλεια των πολιτών. Δεύτερον, Μέσω της ύπαρξης αυτής της δυνατότητας από οποιοδήποτε άλλο προξενείο υπογραμμίζουμε την διάσταση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τρίτον χαιρετίζουμε το ότι η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει μια επικαιροποίηση των διαδικασιών χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων. Πράγματι η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες τροποποιήσεις τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προξενική προστασία και δεν λαμβάνει υπόψη τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι λοιπόν προστατεύει ανεπαρκώς από απάτες και παραχαράξεις και γι' αυτό Υποστηρίζουμε λοιπόν τις προτάσεις ενίσχυσης της ασφάλειάς του. Και τέλος συμμεριζόμεθα πλήρως την άποψη της εισηγητρίας κυρίας Γκάλ και θέλουμε η πρότασή της να γίνει δεκτή χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλέρο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλα όσα θα ήθελα ήδη να πω. Να πω λοιπόν ότι εγώ θα συμφωνήσω με τις προτάσεις. Είναι κάτι το ιδιαίτερο θετικό για τον Ευρωπαίο πολίτη και είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πρέπει να το ενισχύσουμε και εμείς. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της προτάσεως αυτής, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ θετική πρόταση, δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες και θα υποστηρίξουμε την πρόταση ως έχει. Ευχαριστώ, θα ήθελα τέλος να ζητήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στάλλερ Μόσχαμερ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδης. Είναι ένα σημαντικότατο μέσο για τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν έκτατες καταστάσεις στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το 60% των περιπτώσεων που ζητούν προστασία αναφέρεται στην επανέκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου αυτό λοιπόν θα καταστήσει ευκολότερη τη ζωή των ταξιδιωτών και θα διασφαλίσει καλύτερα και την ασφάλειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάλ πάλι. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. για να αποδείξουμε και εμείς από την πλευρά μας ότι είναι πραγματικά ένα θέμα πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου. Άλλαξε η ημερομηνία. Okay, now We start the point number 12. Uh, Ωραία, περνάμε στο 12. Στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνέρων, η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία μια νέα, μιας νέας ε, χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνιακών ελέγχων. Έχουμε γνωμοδότηση. Ο κύριος Λέναρς είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης αυτής και αυτή θα συζητήσουμε τώρα. Θα εξετάσουμε, όπως είπα, το σχέδιο γνωμοδότησης. Σήμερα, λόγω του χρονοδιαγράμματος της ε, ε, ΙΜΚΟ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια ε, επιτροπή, οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις θα γίνουν αποκλειστικά στα αγγλικά. Κύριε Λέναρ, έχετε δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Να τρέξω λοιπόν. Ναι, το συζητήσαμε και όταν παρουσίασε στην Επιτροπή μα την πρόταση η Κομισιόν. Ούτε τότε βέβαια είχαμε πολύ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει είναι, ε, είναι περίπλοκο το θέμα. Είναι νέο ταμείο που ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη. Αποτελεί καινούριο στοιχείο, σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση τη προστασία των εξωτερικών των κοινών μα ε, συνόρων. Γνωρίζουμε ότι οι εγκληματίε γνωρίζουν ποια είναι τα δύναμα στοιχεία σημεία στα σύνορά μας, στα τελωνία μας και προσπαθούμε βεβαίω να τα εκμεταλλεύονται. Άρα είναι καλή πρωτοβουλία η δημιουργία αυτού του ταμείου. Έχω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη δική μου γνωμοδότηση. Πρώτον, όπως είπες σωστά, εντάσσεται στην, ε, στο Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των θεωρήσεων. Έχουν κοινού στόχου, αλλά έχουν και εξειδικευμένου ξεχωριστού στόχου τα, τα δύο ταμεία αυτά και χρειάζεται και από πλευρά Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει επικάλυψη των ταμείων με, όσον αφορά του ε, ε, ειδικού στόχου που εξυπηρετούν, καθώ και στα χρήματα βεβαίω με τα οποία ε, περικοδοτούνται τα ταμεία αυτά. Προσπαθώ λοιπόν να οριοθετήσω καλύτερα με τις ε, τροπολογίες μου α, ε, αυτε, αυτούς τους διαφορετικούς στόχους. Επίσης, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και την Ευρωπαϊκή συνοριοφυλική και Ακτοφυλακή. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να, να σε αυτό το ταμείο. Είναι ένα ταμείο το οποίο θα ενισχύει την ε, διοργανική ε, συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων και εθνικών φορέων, καθώς και του εξοπλισμού που αποκτάται μέσω αυτής της χρηματοδοτικής στήριξης. Επίσης προβλέπεται και αντίστοιχο ε, για το ποιο ε, εξοπλισμός θα ε, αγοραστεί, ποιο θα, θα έχει ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τέλος, η πρόταση επιτρέπει την, την χρήση του εξοπλισμού των ελληνικών ελέγχων για του συνοριακού ελέγχου, υπό, υπό το άρθρο 6 παράγραφο 4. Νομίζω ότι πρέπει να αποσαφινιστεί. Ε, έχω υποβάλει κάποιε προτάσει για τη βελτίωση του, του κειμένου αυτού. Αυτά μπορούσα να κάνω σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω να υπάρχουν σκιώδει, ούτε κάποιο άλλο που να θέλει το λόγο. Αν δεν υπάρχουν σκιώδει, ίσω θα μπορούσα να προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, Έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θέλετε το λόγο, σας παρακαλώ. I'll Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε για την γνωμοδότηση. Την εκτιμούμε. Εκτιμούμε την υποστήριξη για το πρόγραμμα. Ουδέν άλλο σχόλιο. Yeah. Thank you. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε, Κυρίε Λενάς. και αυτό το σημείο. Δεν χρειάζεται να συνοψίσετε αυτή τη συζήτηση. Τώρα ποιο πρόβλημα έχουμε. Δεν έχουμε εδώ τον εισηγητή για το επόμενο σημείο. Then one, two minutes break. Θα σταματήσουμε για ένα-δύο λεπτά.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 προς όφελος των τελικών χρηστών και δικαιούχων. Να σας υπενθυμίσω ότι λόγω του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής Ρέτζη οι συντονιστές πήραν τις αποφάσεις για τον χρονισμό τον οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω την τσεχική. γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη γλώσσα μου, είναι μια ωραία γλώσσα με πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γενικά αποδεκτή θα έλεγα. Προτείνουμε και εμείς κάποιες αλλαγές βέβαια και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε τρεις βασικά τομείς Θέλουμε κάποιους ενιοποιημένους κανόνες, θέλουμε να εναρμονίσουμε επίσης τον τρόπο χρηματοδότησης. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια ικανοποιητική λύση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα χρηματοδότησης, ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σχόλιο των μελών του Κοινοβουλίου, το οποίο έχουμε, έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, εκεί όπου διαπιστώνονται ε, ε, διπλές χρηματοδοτήσεις, υπάρχει δηλαδή πιθανότητα κατάχρησης των ε, κανόνων, η προσοχή μας θα πρέπει να είναι αυξημένη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την νομοθεσία όσο πιο απλή γίνεται. Νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας μπορεί πλέον να γίνει δεκτό. Το οποίο παρέχει το σχέδιο αυτό όλες τις πληροφορίες για τις πηγές χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για την καλή δουλειά την οποία έχουμε κάνει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Ντάλη, σκιώδη εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή. Είναι τυχερός που μπορεί να χρησιμοποιήσει την ωραία του γλώσσα, ενώ δυστυχώς η δική μου ωραία γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη σήμερα. Εν πάση περιπτώσει τον ευχαριστώ για την πολύ καλή του δουλειά. Στηρίζω την προσπάθεια την οποία κάνει και στα πλαίσια των, του κανονισμού κοινών διατάξεων και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο και την μετανάστευση. Εγώ θέλω να τροποποιήσω τον τίτλο και να ενισχύσω τον στόχο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και Γι' αυτό ε, υποστηρίζω τις προτάσεις Βιτσόφσκη των CPI σχετικά με τις προτάσεις του. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Είναι επίσης θετικό ότι γίνεται αναφορά στην χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλα τα κοινοτικά όργανα και θα και μάλιστα αντικατοπτρίζεται και στη δική μου έκθεση σε σχέση με το καταπίστευμα για την μετανάστευση. Εμείς προτείνουμε να καταστήσουμε λοιπόν πιο ευέλικτη την κατανομή των πιστώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες που υπάρχουν στις διάφορες χώρες και απαιτείται εδώ μεγαλύτερη διαφάνεια Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι στον εισηγητή, κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Η κατεξουσιοδότηση πράξης για τα εθνικά προγράμματα ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε. είτε στην παρούσα φάση είτε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει το λόγο. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος που θα, θέλα, θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι κανένας από όλους αυτούς που είπατε. Ούτε ο κύριος Βαλίλα, ούτε ο κύριος Τευτευτριάγια, ούτε Φατσινέλο. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, για τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική του στάση. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να εναρμονίσουμε τις ε, προσεγγίσεις με τα ταμεία κοινή διαχείρισης για να ε, προσφέρουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα διέπουν τα ταμεία αυτά και θα απλοποιούν τη ζωή ε, θα διευκολύνει τη ζωή των ε, κρατών μελών, των αρχών, των δικαιούχων και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και με αυτόν τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Παρ' όλα αυτά βεβαίω, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για τις προτάσεις που κάνει για την απλοποίηση του κειμένου. Υπάρχουν μια σειρά από προτάσει του που πραγματικά αποσαφηνίζουν αυτό και που και εμείς προσπαθούσαμε να πούμε για τα, τα τρία βασικά ταμεία ιδίω ε, θεωρούμε ότι είναι αξιέπινη η προσπάθεια, η προσπάθειά του να ληφθούν υπόψη κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Να εξηγήσω λίγο το σκεπτικό από πλευράς Κομισιόν. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι για τον τίτλο του Ταμείου ε, Ασύλου και Μετανάστευσης. Σκόπος της Κομισιόν με την αλλαγή του ονόματος ήταν στην, πραγματικά, πραγματικότητα η απλοποίηση. Γιατί η μετανάστευση ε, περιλαμβάνει και την κοινωνική ένταξη και συνολικά τα ζητήματα ε, των, ε, ε, της μετανάστευσης. Δεν ήταν απλώς ο σκοπός μας να μειώσουμε τις λέξεις του τίτλου, αλλά να ε, είμαστε πιο ευσύνοπτοι. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που προτείνει ο σχετικά με τις παρατηρήσεις της Κομισιόν για τα περιφερειακά προγράμματα και τα εθνικά προγράμματα. Εδώ να σας πω ότι η διατύπωση που είχαμε επιλέξει την επιλέξαμε με πολύ προσεκτικό τρόπο. Μπορώ να σας εξηγήσω και διμερώς ποιο ακριβώς ήταν το σκεπτικό μας. Αυτό που θέλαμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός ίσχυε μέχρι στιγμής χρειαζόταν η Κομισιόν, παρόλο που δεν, δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση όταν θεσπίστηκε, να υποβάλει έκθεση υποχρεωτική για τις παρατηρήσεις της. Δηλαδή διπλασιαζόταν το έργο. Αυτό που λέμε τώρα πλέον είναι δεν χρειάζεται επίσημη απόφαση για τις παρατηρήσεις και να αντικατασταθεί αυτή η διαδικασία με, τις, με την ανταλλαγή επιστολών, με την αλληλογραφία, κάτι που θα επιταχύνει συνολικά τις διαδικασίες, θεωρούμε. Οι τροπολογίες που σχετίζονται με τις προθεσμίες της Κομισιόν, η εξήγηση από πλευρά μας εδώ είναι ότι έχουμε ε, διδαχθεί από την προηγούμενη περίοδο και το βασικό δίδαγμα είναι ότι οι, οι τρέχουσες ε, προθεσμίες, οι ισχύουσε προθεσμίε, είναι πάρα πάρα πολύ στενέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο χρόνο, το αναγνωρίζουμε αυτό, χρειαζόμαστε να έχουμε στη διάθεσή μα τον επαρκή χρόνο για να μπορούμε να αναλύουμε τα προγράμματα, να ανταλλάσσουμε απόψει και πληροφορίε με τα κράτη-μέλη και να οριστικοποιούμε στη συνέχεια τις θέσεις μα. Και τελικό σημείο που σχετίζεται με μία από τι τροπολογίε για την εισαγωγή της έννοιας των ε, εμβληματικών προγραμμάτων. Νομίζω ότι ιδίω σε σχέση με κάποια τουλάχιστον ταμεία, τι να σα πω, σημειώνουμε την ιδέα σας αυτή, ε, μας ενδιαφέρει και εμάς η ορατότητα και η προβολή των προγραμμάτων, μια ανησυχία που ίσως έχουμε είναι ότι η έννοια αυτή δεν ορίζεται πουθενά αλλού στον κανονισμό. Σω θα πρέπει λοιπόν να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο ορισμό προκειμένου να ξεκαθαρίζονται και οι επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη για το πώ ακριβώ θα, θα λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη και ποια καθήκοντα βεβαίω θα συνεπάγεται ε, ε, ένα τέτοιο χαρακτηρισμό ω εμβληματικού προγράμματο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Μίριαμ. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ για τα σχόλια. Τα σημειώνω όλα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, θα καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας. Και θέλω να ξανατονίσω ότι η πρότασή σας ήταν εξαιρετική, καθόλου εξαιρετική. Απλώς εγώ προσπαθώ να βελτιώσω κάποιες λεπτομέρειες που κατά τη γνώμη μου δεν είναι απολύτως σαφείς. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να κάνουμε κάποιες διμερείς επαφές, ώστε το κείμενο να είναι απόλυτα σαφές σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλους τους αναγνώστες. Δεν θα, δεν θα περιλαμβάνει ούτε σφάλματα, ούτε παρεξηγήσεις. Να έχουν όλοι ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς προβλέπετε. Είμαι ανοιχτό στο διάλογο βεβαίως μαζί σας και είμαι βέβαιος ότι από κοινού θα καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι προς όφελος και δικό μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πρόεδρος. Ωραία. Έχουμε 10 λεπτά μέχρι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το σημείο 14. Because as I understand... Aha, yes, sorry. Sorry. Α, με συγχωρείτε. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 24 Οκτωβρίου. Έγκριση της γνωμοδότησης 21 Νοεμβρίου. Αλλά τροπολογία σε μια πρώτη φάση είπαμε 24 Οκτωβρίου. 6 το απόγευμα. Λοιπόν, όπως έλεγα, θα κάνουμε ένα δεκάλυπο διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. 11.30 ακριβώς.